Ε, σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη πρέπει να εξετάσουμε την κατάσταση στο Αζερβαϊτζάν και το λόγο έχει η κυρία Λούνατσεκ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, Επίτροπε, κυρίες και κύριοι. Στην Ανατολική γειτονία, δυστυχώ, το Αζερβαϊτζάν έχει μετατραπεί σε μια χώρα που έχει τι χειρότερε επιδόσει στα ανθρώπινα δικαιώματα. Ακόμα και η Λευκορωσία πρόσφατα απο, ε, αποδέσμευσε, αποφυλάκησε έξι πολιτικού κρατημένου. Πρέπει λοιπόν τα ανθρώπινα δικαιώματα να βρίσκονται και είναι στο επίκεντρο των σχέσεων τη Ευρωπαϊκή Ένωση με τρίτε χώρε και πρέπει ενωμένοι να αγωνιστούμε δίπλα σε αυτού που προσπαθούν να φέρουν τα ανθρώπινα δικαιώματα του κράτου δικαίου και τη δημοκρατία τη χώρα. Δεν μπορούμε να έχουμε δίπλα μέτρα και σταθμά για μας και για του άλλου. Πρέπει λοιπόν να καλέσουμε, για, να απευθύνουμε έκκληση για την ε, μέση αποφυλάκηση όλων των πολιτικών ε, κρατουμένων, να εκφράσουμε την ικανοποίησή μας για την άδεια για επίσκεψη στην ε, στους ε, κρατημένους στη Λεϊλά και τον Αρίφ και ελπίζω, κλείνοντας να πω ότι ελπίζω να με παρακολουθούν και οι αρχές του Αζερβαϊτζάν γιατί ζητεί το ψήφισμα μας να τηρηθούν όλες οι αποφάσεις του Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων συμπεριλαμβανομένης και αυτής της Δευτέρας Ιουνίου του 2015 όπου καταγγέλλεται η παρουσία και η κατοχή από πλευράς της Αρμενίας εδαφών του Αζερβαϊτζάν. Ευχαριστώ πολύ. Κύριο Καρίμ, Πρόεδρε ευχαριστώ και ξεκινώ με ένα απόσπασμα από μια παλαιά ομιλία που εκφωνήθηκε πριν από 40 χρόνια στο Στρασβούργο το Αζερβαϊτζάν έχει πάρει, πριν από 14 χρόνια, συγγνώμη, ε, το Αζερβαϊτζάν έχει πάρει το δρόμο για το κράτος δικαίου, τη δημοκρατία και τις ανθρώπινες αξίες. Ο Χάιντερ Αλιεύ το 2001 εκφώνησε το λόγο αυτό εδώ. Και όμως μια ιστορία απογοητεύσεων ήταν αυτή του Αζερβαϊτζάν και μάλιστα θα έλεγα και αμοιβαίων απογοητεύσεων για να είμαστε ειλικρινεί. Επί παραδείγματι γνωρίζουμε ότι το Αζερβαϊτζάν αισθάνεται δυσφορία σε σχέση με την απουσία πρόοδο στην υπόθεση του Ραγκόρνο Καραμπάχ. Ξέρουμε επίση ότι θεωρεί πω η διεθνή κοινότητα αγνοεί τι μεγάλε προκλήσει με τι οποίε βρίσκεται αντιμέτωπο ύστερα από τον πόλεμο αυτόν σε σχέση με του πρόσφυγε, σε σχέση με του εσωτερικά Και Όντω δεν έχει επιδείξει την ενεργητικότητα που θα όφιλε η διεθνή κοινότητα για να ε, αντιμετωπίζει για να αντιμετωπίσει αυτήν την ε, σύγκρουση, η οποία πρέπει να το πούμε, αλλά δύο λάθη δεν ισοδυναμούν με ένα σωστό και πρέπει και να τηρηθούν οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Ανθρωπινών Δικαιωμάτων για τα εις των ανθρωπινών δικαιωμάτων που γεννούν πολύ σοβαρές ανησυχίες όπως διαπιστώνεται η κατάσταση σήμερα για να το πω διπλωματικά. Και θα ήθελα επίσης να σημειώσω ότι επί της αρχής είναι σαφές, είναι απλά τα πράγματα. Το Αζερβαϊτζάν πρέπει να ξαναβρει το δρόμο του προς ένα ευρωπαϊκό μέλλον. Ευχαριστώ. Αξιότιμοι συνάδελφοι, σας παρακαλώ να τηρείτε το χρόνο που σας έχει δοθεί. Γιατί αν μιλάτε περισσότερο χρόνο, κλέβετε το χρόνο από τους συναδέλφους που έχουν ζητήσει να παρέχουν το ΚΑΤΣΙΑΙ. Στις 12 πρέπει να ψηφίσουμε, οπότε λάβετε υπόψη τι, το τι κάνετε απέναντι στους δικούς σας συναδέλφους. Ο κύριος Πρέντα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εξ ονόματος του ΕΛΚΟ θα ήθελα να πω δύο πράγματα. Καταρχήν εκφράσαμε στο ψήφισμά μας ε, την ανησυχία μας ε, σε σχέση με την κατάσταση της υγείας της Λέιλα και του Αρήφ Γιούνους και εκφράζουμε την επιθυμία μας να απελευθερωθούν όσο γίνεται πιο σύντομα. Η σιωπηρή διπλωματία είμαστε ικανοποιημένοι που έφερε αποτελέσματα γιατί μπορέσαμε να του βοηθήσουμε τουλάχιστον από ιατρική άποψη. Απ' την άλλη πλευρά δεν ψηφίσαμε, δεν, το κοινό, δεν υπογράψαμε συγγνώμη, το κοινό ψήφισμα γιατί δεν στηρίζουμε την στρατηγική των Πρασίνων, δηλαδή να ερχόμαστε στην Ολομέλεια χωρί να περνάμε από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και να ζητάμε από την Ολομέλεια να αποφασίσει για τα μέσα τη πολιτική γυρνίασης ε, για τις έρευνες που γίνονται από το θεσμού της Ένωσης για τον πρόεδρο Αλιέφ που είχε συνυπογράψει με τον πρόεδρο Τούσκ ε, ε, συμφωνίες για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και στον τομέα του δικαίου. Αυτή η στρατηγική των πρασίνων δεν είναι σωστή, δεν τη δεχόμαστε και θα ζητήσουμε μάλιστα να μην γίνει ψηφοφορία για αυτό το ψήφισμα σήμερα, γιατί αποδεικνύει έναν ριζοσπαστισμό που δεν έχει παρά μόνο τα αντίθετα αποτελέσματα. Ο κύριος Κοράου. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είναι αλήθεια, λίγο τυχαία, λίγο κατά σύμπτωση. Σε αυτή τη σύνοδο ε, μιλήσαμε και τόσο για τη Λευκορωσία όσο και για το Αζερβαϊτζάν. Και είναι πολύ ωραίο να βλέπουμε πώ αυτό το κοινοβούλιο ε, προσεγγίζει με διαφορετικά μέτρα και σταθμά δύο χώρε που γεωγραφικά ανήκουν στην ίδια περιοχή και που μπορούν να τοποθετηθούν σε μια ταξινόμηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αν θέλουμε να κάνουμε τέτοιου είδου ταξινόμηση, εν πάση περιπτώσει, μάλλον οι παραβιάσει στα Αζερβαϊτζάν είναι χειρότερε από αυτέ στη Λευκορωσία. Όμω στη Λευκορωσία βάζουμε ε, κυρώσεις, ενώ στο Αζερβαϊτζάν κάνουμε business. Γιατί είναι σαφές ότι η λογική αυτής της στρατηγικής, την οποία μόλις ε, ε, ανέφερε και ο συνάδελφος Πρέντα, το Αζερβαϊτζάν μας χρησιμεύει γιατί μας δίνει υδρογονάνθρακες και δεν θέλουμε να εξαρτάμαστε μόνο από τη Ρουσία. Οπότε τι μα νοιάζει άμα το Αζερβαϊτζάν παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα, άμα βασανίζει ε, δημοσιογράφους. Το χρησιματικό είναι να κάνουμε business. Τελείω λάθο αυτό το είδους η στάση την οποία κρατά το ΕΛΚ που δεν θέλει καν να την ψηφίσουμε γιατί άμα είναι έτσι ε, να βάλουμε ε, καλύτερα να βάλουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα πριν από τα business που θέλουμε να κάνουμε με το Αζερβαϊτζάν και να την ψηφίσουμε σήμερα το ψήφισμα. Μπορεί να μην ε, αρέσει στον ε, κύριο Πρέντα. Το Κοινοβούλιο εδώ και ε, μήνε καταγγέλει με την κατάσταση στο Αζερμπαϊτζάν. Η Κομισιόν πρόσφατα είπε ότι έχει επιδεινωθεί σημαντικά η κατάσταση των ανθρωπινών δικαιωμάτων ε, στη χώρα. Υπάρχει συμφωνία σύνδεση με το Αζερμπαϊτζάν και η σύμβαση σύνδεση είναι κάτι το οποίο, για το οποίο πιέζει το Συμβούλιο και το ε, και η Κομισιόν. Ε, τον Ιούλιο ε, θα πάει να επισκεφθεί τον κύριο Αλίεφ, τον κύριο Στούσκα. Α, όχι κύριε Πρέντα, δεν ενορχιστρώνουμε, τα χειραγωγούμε εμεί τα πράγματα και δεν είστε και σε καλή θέση για να δίνετε και σε εμά μαθήματα. Σταματήστε λοιπόν. Έχουμε τις σχέσεις με τη Ρωσία. Έχουμε και τον ορυκτό πλούτο της χώρας. Ίσως αυτά να εξηγούν και τη στάση των δύο θεσμικών οργάνων της Ένωσης και τη δική σας, ε, κύριε Πέντα. Πώς μπορούμε να είμαστε αξιόπιστοι για να αποφύγουμε για μια ακόμη φορά να θυσιαστούν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δύο μέτρα και δύο σταθμά εξηγούν αυτά το φαινόμενο της ατιμορρησίας ε, της ε, κυβέρνησης της χώρας αυτής που καταστέλει τους ακτιβιστές που ε, θέλουν, που την χάνουν του άκρα του σεβασμού. Σε κυρία Σάκε, έχουμε συστηματικές παραβιάσει των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, στο Αζερμπαϊτζάν, Ισμαήλοβα, η Λέλα Γιούνουσε, ο Αρίφ Γιούνουσε έχουν καταδικαστεί σε εξωφρενικές ποινές, αλλά και πολλοί άλλοι ακτιβιστές, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημοσιογράφοι, οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών αντιμετωπίζουν καταστολή, βία, και αυτοί που ζητούν τώρα περισσότερο χρόνο για τη σιωπηρή διπλωματία, τι να πω, οι Αζέροι, ε, οι Αζέρικες αρχές είχαν όλο το χρόνο στη διάθεσή τους για να ε, φροντίσουν να γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα και να τηρούν και τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει ότι θα εφαρμόσουν τις αποφάσεις ε, του, Συμβουλίου, του Δικαστήριου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ε, και τις εστάσεις ε, του ΑΣΕ. Σεβασμό της δημοκρατίας, σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν μας χρειάζεται ένα είδους ρωσικού σενάριου αυτή τη φορά στο Αζερμπαϊτζάν. Πρέπει λοιπόν να μιλήσουμε τώρα και να πούμε ποια είναι η εναλλακτική βλέποντας τόσο σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τι μπορεί να πετύχει η ισοπηρή ε, διπλωματία. Ναι, καλός είναι ο διάλογος, αλλά με ηχερά μηνύματα. Και μέχρι τώρα έχουμε δει οι ισοπηρέ μας προσπάθειες να μην αποδίδουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Κύριε πρόεδρε, δεν μας απασχολεί για πρώτη φορά. Το Αζερβαϊτζάν είναι πάγιος προσκεκλημένος των συζητήσεών μας. Θέλει να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση με μεγάλες ε, εκδηλώσεις, οργάνωσε ζήτησε μάλλον Ολυμπιακούς Αγώνες. Ε, είναι κάτι όμως το οποίο βλέπουμε να αφήνει πάρα πολλά κενά ως προς την τήρηση των συνθήκων του κράτους δικαίου, το σεβασμό των ανθρωπινών δικαιωμάτων έχουμε δικαίωμα να ρωτάμε, γιατί είναι και μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης και έχει συνυπογράψει την Επιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, τη Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, βλέπουμε ότι παραβιάζει και αγνοεί κάθε έννοια δικαίου και δημοκρατίας. Δεν είναι επιφανειακά σχόλια αυτά. Είναι σοβαρή η κατάσταση και δεν μπορούμε να παρετηθούμε από την επιδίωξη τη επιβολή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Αζερβαϊτζάν, αλλά και προ όφελο και του ευρωπαϊκού συμφέροντο, όχι μόνο για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Αζερβαϊτζάν. Ευχαριστώ πολύ. Τουν und Holstein. Πρόεδρε, στη χώρα του Αλίεφ Έχουμε διπλάσιο αριθμό πολιτικών κρατουμένων σήμερα από ότι στη Ρωσία και τη Λευκορωσία μαζί. Οι συνθήκες οι οποίες κρατούνται είναι γνωστές. Δεν φαίνεται όμως να ενδιαφέρεται ο πρόεδρος του Αζερβαϊτζάν ούτε για ανθρώπινα δικαιώματα ούτε για διεθνείς δεσμεύσεις. Αυτό απαιτεί να εκφράσουμε εμείς με απερίφραστο τρόπο τις θέσεις και τις απαιτήσει μας. Θυμόμαστε πολύ καλά την εποχή που ζούσαμε κάτω από τη δικτατορία, κάτω από τον κομμουνισμό, που αγωνιζόμασταν για αυτά τα δικαιώματα. Και τότε μας είχε προσφερθεί υποστήριξη, ευρεία υποστήριξη και με ε, δηλώσεις και με εμπλοκή πρακτική του Ευρωπαϊκού, Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλων ε, και άλλων ε, θεσμών. Λυπούμε λοιπόν που η ομάδα μου, η πολιτική, δεν έχει προσυπογράψει το ψήφισμα αυτό. Για τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν είναι ζήτημα πολιτικής, πολιτικού προσανατολισμού. Είναι απόλυτα. Και καλό την ομάδα μου να υπερψηφίσει το ψήφισμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πύρη. Πύρη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πριν από ένα χρόνο μιλούσαμε για τα ίδια πράγματα, για την σύλληψη ακτιβιστών ε, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημοσιογράφων και δικηγόρων του Αζερβαϊτζάν. Πρόεδρε, εσείς ε, είπατε για τη Λέιλα Γιούνους και προπορτάθηκε για το βραβείο Ζαχάροφ και παρότι το Αζερβαϊτζάν είναι σημαντική χώρα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι επικρίσεις μας δεν έφεραν κανένα αποτέλεσμα. Μετέβαινε εκεί το περασμένο καλοκαίρι, κυρίως και μάλιστα μετά από ότι την ε, δίκη τη κυρία Γιούνους και του συζύγου τη. Βρίσκονται μέσα σε ένα γυάλινο κλουβί, δεν μπορούσαν να συζητήσουν καν με δικηγόρο. Ο Αλέφη Γιούνουφ χρειάζεται να μεταφερθεί με νοσοκομείο στη διάρκεια της δίκης, γιατί υπεφέρουν ε, από διάφορες ε, ασθένειες μετά το πέρας της δίκης ε, καταδικάστηκαν σε 6-7 χρόνια φυλάκισης έκαστος, δηλαδή καταδίκη σε θάνατο στην ουσία. Δεν είναι δυνατόν οι διπλωματικές υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι Κομισιόν μέχρι στιγμής να μην έχουν παρέμβει πιο σταθερά και πιο έντονα απέναντι σε αυτή την κατάσταση στο Αζερβαϊτζάν. Η καταδίκη αυτή και, ε, ε, της Λέιλα και του Αρίφ είναι εφικτή και η κυρία Ισμαήλοβα και ο κύριο Αλιέφ είναι αθώοι που βρίσκονται στην ε, φυλακή. Πρέπει να τους ζητήσουμε άμεση απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων. Σημαντικό κομμάτι της πολιτικής γυρνίας τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η πολιτική περισσότερα για περισσότερα. Όσε περισσότερε μεταρρυθμίσει γίνουν, τόσο περισσότερη βοήθεια θα δοθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το αντίθετο θα έπρεπε να ισχύει όμω, λιγότερα για λιγότερα. Ζητάμε από το Αζερβαϊτζάν να, να τηρήσει τι υποχρεώσει του ω μέλο του Συμβουλίου τη Ευρώπη ε, και μέχρι στιγμή η ομάδα μου ζητά να υπάρξουν και στοχευμένε ε, οικονομικέ κυρώσει καθώ και η πάυση τη χορήγηση βίζα ε, σε όσου αναμειγνύονται σε πολιτικέ διώξει. Βάγγελ, Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπη, κύριε Πρόεδρε. Κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ε, του κράτο δικαίου, ιδίω σε χώρε με τι οποίε έχουμε συμφωνίε εταιρική σχέση ε, και μπορούμε να επικοινωνούμε μαζί του, ε, είναι ένα θέμα το οποίο μα απασχολεί ιδιαίτερα στο Κοινοβούλιο και το Αζερμπαϊτζάν είναι πολύ συχνά στη μερίσια διάταξη των εργασιών του Κοινοβουλίου. Συζητούμε ένα πολύ σκληρό ψήφισμα σήμερα και έχουμε καλού λόγου γι' αυτό. Ελπίζουμε να έχει θετικό αντίκτυπο το ψήφισμά μα, φοβούμε ότι δεν θα έχει. πολλές φορές ε, ε, θεωρεί το Αζερβαϊτζάν ότι επικρίνεται πολύ περισσότερο από ότι γειτονικέ χώρες ε, όπως είναι η Αρμενία για παράδειγμα έχουμε το θέμα του Ναγκόρνο Καραμπάχ, έχουμε το 3% που κατέχεται παρουσία ρωσικού στρατού κτλ. Είναι μια χώρα που πρέπει να προσέξουμε, πρέπει να της ασκήσουμε κριτική, αλλά πρέπει να δούμε και την όλη περιοχή. Ευχαριστώ πολύ. Για μια ακόμη φορά συζητούμε τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Αζερμπάιτζαν. Το 2009 το Κοινοβούλιο ήδη κρίσω τον κόδωνα του κινδύνου ε, για την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων επί αλήφ. Έκτοτε συνεχώς ε, αναφέρουμε αυτή την ε, απολυταρχική εκτροπή, η οποία σοβητή νόημα είχαν όλα αυτά. Το καθιστός Αλίεφ και καταργεί τα θεμελιώδη δικαιώματα, αλλά προσπαθεί να περάσει και τις γειτονικές δημοκρατίες, στρατιωτικές επιθέσεις στην Αρμενία και το θέμα του Ναγκόρνο Καραμπάχ ακόμη ε, δεν έχει επιληθεί. Τη Δευτέρα ε, στο Cash Investigation της France 2 ε, βλέπουμε ότι προσπαθούν να αγοράσουν διεφθαρμένους πολιτικούς ε, δηλαδή βάζουν πλέον το πόδι τους και στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρόλα αυτά είναι τέρος μας αυτή η χώρα πώς αυτό το καθεστώς μπορεί να εκμεταλλεύεται αυτή την πολιτική γειτονία. γιατί είναι ένα καθεστώς που προσπαθεί να υπονομεύσει τις αρχές μας δεν τις υποστηρίζει, δεν τις ενστερνίζεται έχουμε πολλούς κρατουμένους δημοσιογράφους και άλλου ακτιβιστέ. Πρέπει να του υποστηρίξουμε. Ευχαριστώ. μισή λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας εκτιμώ ιδιαίτερα και γι' αυτό θα κάνω το σοβαρό μπονάνο σήμερα. Λοιπόν, όσον αφορά το θέμα του Αζερβαϊτζάν, να πω ότι αισθάνομαι φίλο των Αζέρων και του Αζερβαϊτζάν και δεν συμφωνώ καθόλου με τα όσα άκουσα μέχρι τώρα. Αυτό το επίγον ψήφισμα σε τι χρησιμεύει. Χρησιμεύει στην ουσία όταν κανεί αντί να ε, σκαλίζει τη μύτη του, παίρνει ένα χαρτομάτιλο και φυσάει τη μύτη του εκεί. Δηλαδή, τι ναι, λέμε ότι είναι ε, μας απασχολεί το Αζερβαϊτζάν. Λέμε όμως τίποτα συγκεκριμένο, είναι γελίο. Παράγουμε χαρτί εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο που δεν χρησιμεύει τίποτα άλλο παρά σαν χαρτομάδιλο. Τώρα μιλάτε για το Ισλάμ. Το μετριοπαθές Ισλάμ υπάρχει στο Αζερβαϊτζάν. Υπάρχουν περισσότερα δικαιώματα για τι γυναίκε από ό,τι αλλού. Υπάρχει μετριοπαθές Ισλάμ, ναι ή όχι. Ναι, υπάρχει. Μα όταν λέτε ότι δεν υπάρχουν δικαιώματα, μα τότε αγαπητοί Ευρωπαίοι, γιατί κάνετε business με την Κίνα. Το τελευταίο χρόνο 700 άνθρωποι εκτελέστηκαν εκεί για την Ιγυρία. Εντάξει, εκεί υπάρχει πετρέλαιο, οπότε την Ιγυρία την βλέπουμε με διαφορετικό τρόπο και ούτω καθεξή με όλε τι χώρε Ποια είναι η ουσία. Όπω είπε και πριν κάποιο συνάδελφο δεν είναι ότι κάθε φορά έχουμε άλλα μέτρα και σταθμά. Εκατό διαφορετικά μέτρα και σταθμά έχουμε, όχι μόνο δύο. Εγώ λέω ζήτω λοιπόν τα Αζερβαϊζάν, ζήτω οι Αζέρια, πάμε εκεί και α μιλήσουμε μαζί του σε μια πραγματική στρογγυλή τράπεζα, όχι με τα λόμπι που μεταταλλάζουν. Η Ευρώπη πρέπει να πάει εκεί να, μιλήσει, να, να μαζί τους και να βρει λύσεις. Αυτός είναι ένας σοβαρός τρόπος για μια αξιοπρεπή εξωτερική πολιτική. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Πρόεδρε, συμφωνώ. 100% θα πρέπει να σκεφτεί κάθε δυνατή πίεση στο Αζερβαϊτζάν ώστε να σεβαστεί τα ανθρώπινα δικαιώματα και ακριβώς αυτό είναι το νόημα της σημερινή πρόταση ψηφίσματος. Γι' αυτό λυπούμαστε που το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα βρέθηκε στη θέση, σε θέση να μην υποστηρίζει το ψήφισμα αυτό. Πρέπει να αντλήσουμε όμως τα διδάγματα αυτής της κατάστασης. Πρέπει να προσπαθούμε πάντα το στο Κοινοβούλιο να εκφράζουμε ψηφίσματα τα οποία να είναι ενωτικά και κοινά για όλες τις πολιτικές ομάδες. Για μας η διατύπωση ότι αμέσως, αμέσως είναι η λέξη που χρησιμοποιείται, να διακοπούν οι διαπραγματεύσεις με το Αζερβαϊτζάν θα ήταν μεγάλο λάθος γιατί εάν συμβεί αυτό με όλες τις χώρες του κόσμου θα έχουμε διαπραγματεύσει με κανέναν εν τέλει. Και να ακολουθήσουμε μια τέτοια γραμμή. Αν ακολουθούσαμε μια τέτοια γραμμή με το Ιράν δεν θα είχαμε τώρα πυρηνική, ε, συμφωνία για τα πυρηνικά. Ας κάνουμε λοιπόν το περισσότερο. Ας κάνουμε αυτά που κάνουμε για τη μία χώρα και για την άλλη. Για να μην βρισκόμαστε ενώπιον αυτών των καταστάσεων. Θέλουμε το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Αζερβαϊτζάν, αλλά θέλουμε όλα να γίνουν σωστά. Ευχαριστώ πολύ και τώρα η διαδικασία Καριστιάλ. Παρακαλώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Αζερβαϊτζάν πρέπει να συνεχίσουν τη συνεργασία όπως ε, δήλωσε πρόσφατα και ο πρόεδρος Αλίευ στις Βρυξέλλες στην μια επίσκεψή του. Αυτά λοιπόν που έχουν να κάνουν ε, όχι μόνο με τα ενεργειακά θέματα αλλά και με τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος. Πρέπει να εκφράσουμε απερίφραστα τις ανησυχίες μας για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Αζερβαϊτζάν και ζητούμε από τις αρχές να δώσουν λύση στα προβλήματα και ταυτόχρονα πρέπει να επισημάνουμε ότι τέτοιε ε, καταστάσεις απομακρύνουν τη χώρα όλο και περισσότερο από τη δημοκρατία και τις ανθρώπινες αξίες ε, και τις συμβάσεις τις οποίες έχει ε, προσυπογράψει το Αζερβαϊτζάν. Ταυτόχρονα όμως πρέπει να κρατήσουμε ανοιχτό το διάλογο με το Αζερβαϊτζάν και να ενισχύσουμε την εταιρική σχέση. Αυτό το δρόμο πρέπει να ακολουθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να αποφύγουμε επιλογές που μας μετατρέπουν σε δικαστές και κριτέ, πράγμα το οποίο μα απομακρύνει περισσότερο από το Αζερβαϊτζάν και από τη δυνατότητα διαπραγμάτευση. Ευχαριστώ πολύ. Ο επόμενο ομιλητή δεν είναι στην αίθουσα. Πολύ σημαντική χώρα για την Ευρωπαϊκή Ένωση το Αζερβαϊτζάν. Όμως ε, ε, επειδή επεκτείνει την επιρροή της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τις ανατολικές χώρες και τις ε, έλκει προς εμάς. Ορισμένοι θεωρούν πως η ανατολική εταιρική σχέση είναι ε, για να μπορούμε να πηγαίνουμε να δίνουμε διδά, κηρύγματα, να κάνουμε κηρύγματα στους άλλους. Βεβαίως έχουμε κάποιες ανησυχίες για το τι συμβαίνει στο Αζερβαϊτζάν, αλλά ας μην κάνουμε τους κήρυκες, δεν είναι καλός τρόπος. Ε, τα παραδείγματα είναι που μένουν. Ο Γιάκοπτσιτς ε, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Από το 2009 μέχρι σήμερα το Ευρωκοινοβούλιο έχει οθετήσει 7 ψηφίσματα για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Αζερβαϊτζάν ε, τα στοιχεία για τα οποία μιλήσαμε σήμερα στη διάρκεια αυτής της συζήτησης αποδεικνύουν πως, δεν υπήρξαν, ε, πως υπήρξαν 7 ψηφίσματα, όχι μόνο ένα. Ε, το ελευθεροκτόνο αυτό καθεστώς έχει καταργήσει κάθε μορφή δημοκρατίας στο Αζερβαϊτζάν και δεν είναι και μυστικό ότι οι συνεχιζόμενοι βομβαρδισμοί συνεχίζονται από τη, στις όμορες χώρες, στην Αρμενία, στον ακόρνου Καραμπάκ από την, ε, το καθεστώς ε, του, του Αζερβαϊτζάν. Ε, καθήκον μας είναι να υιοθετήσουμε αυτό το ψήφισμα ακόμα για το, το 8ο ψήφισμα, όχι μόνο γιατί όσα έχουν υιοθετηθεί από το 2000 να, να, γίνουν, να μπουν στη πράξη, αλλά για να αποκατασταθεί μια δημοκρατία για το λαό των Αζέρων, γιατί αυτοί αξίζουν τη δημοκρατία ε, το καθεστώς όμως της χώρας αξίζει μόνο κυρώσεις που θα επιστρέψουν την ελευθερία στον κόσμο. Πώς πιζίλ. Δεν είναι στην αίθουσα. Α, είναι, είναι. Ευχαριστώ. Παρακολουθώ με πολύ προσοχή τη συζήτηση. Ένα από τους συναδέλφους ε, είπε τι νόημα έχει ένα ψήφισμα εφόσον η κατάσταση στο Αζερβαϊτζάν δεν αλλάζει. Διαφωνώ. Ένα ψήφισμα το οποίο καταδικάζει την αδικία στο Αζερβαϊτζάν είναι ένα λογικό ψήφισμα γιατί είναι ένα μήνυμα ε, της στήριξής μας για την αντιπολίτευση. Είναι μια ηθική υποστήριξη Δημοσιογράφος Χαντίτσα Ισμαήλ. 7,5 χρόνια ε, κάθυρξη είναι η ποινή στην οποία καταδικάστηκε μετά από μια άδικη δίκη ε, προσφάτως. Πρέπει να ακουστούν αυτά τα πράγματα και πρέπει ε, να δηλώσουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση την υποστήριξή μας προς αυτούς τους ανθρώπους. Παρακολουθούν, η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί την κατάσταση και οι άνθρωποι αυτοί είναι στραμμένοι σε εμά. Έχουν τις ελπίδες μας και στους αρνές και δεν είναι πάρω. Μια λόβα. Ε, EUn tulee kaikissa tilanteissa puolustaa ihmisoikeuksia ja... Σε κάθε περίσταση θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να προασπίσει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και συμφωνώ με τους ε, συναδέλφους που υπογράφουμε το ψήφισμα. Έχει επιδεινωθεί η κατάσταση στο Αζερβαϊτζάρας προς τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το ψήφισμα πάντως ζητεί επιβολή κυρώσεων, ζητεί πάγωμα της πολιτικής ε, γειτονίας, ζητεί να τηρηθούν ορισμένοι όροι. Πρόκειται για ζητήματα τα οποία πρώτα θα έπρεπε να έχουμε συζητήσει και προετοιμάσει στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Δεν πρέπει να βρεθισκόμαστε εδώ ενώπιον ενός ε, εγγράφου το οποίο έχουν αποφασίσει κάποιοι και κεκλεισμένων των θυρών. Χρειάζεται σωστή προετοιμασία για τέτοιου τύπου ψηφίσματα. Ένα ψήφισμα με σωστή προετοιμασία θα μας δώσει τα αποτελέσματα που θέλουμε. Αλλά όχι αυτό, το οποίο μπορεί να οικονοποιεί ορισμένου, αλλά εμείς πρέπει να επικεντρωθούμε στο γεγονός ότι χρειάζεται να προαχθούν αποτελεσματικά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να καταδικάσω, λέει ο κ. Πόλτσακ, αυτή την συγκεκριμένη υπόθεση και άλλες μας έχουν απασχολήσει. Τα ανθρώπινα δικαιώματα ποτέ δεν θα πρέπει ε, να αντιμετωπίζονται διαφορετικά ανάλογα με τη χώρα Καλό την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους φορείς της ε, να δουν κατά πόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσαν να ληφθούν υπόψη οι διεθνείς αποφάσεις, ε, ε, η τελεσή της αποφάσεις των διεθνών δικαστηρίων. Έχουμε και τις αποφάσεις του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Στρασβούργου. ένα συνάδελφος ρώτησε τι θα σκεφτεί το Αζερβαϊτζάν ε, με αυτό το ψήφισμα. Ναι, είναι προφανέ ότι μπορεί και να μην φέρει κάποιο αποτέλεσμα το ψήφισμα. Αν βρούμε όμω ω Ένωση έναν τρόπο να επιβάλλουμε το κράτο δικαίωμα τη δημοκρατία, ίσω είναι καλό αυτό. Κύριο Μαριά. Κύριε Πρόεδρε, τον Ιούνιο πριν από του Ευρωπαϊκού Αγώνε, για καθαρά πολιτικού λόγου και σκοπιμότητε, έγινε συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το Αζερβαϊτζάν. Τώρα και εν ώψη των κοινοβουλευτικών εκλογών του Νοεμβρίου του 2015 έχουμε κατάθεση ενός νέου πολιτικά φορτισμένου ψηφίσματος ενός ψηφίσματος που δεν είναι ισορροπημένο είναι μονομερές και με συγκεκριμένη πολιτική στόχευση. δυστυχώς το ίδιο το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο μπήκε σε λάθος ατραπούς αφού αποφάσισε να μην στείλει καν παρατηρητές κατά τη διεξαγωγή των κοινοβουλευτικών εκλογών του νοεμβρίου. η τακτική απομόνωση του αζερμπαϊτζάν είναι λανθασμένη οδηγεί σε απομόνωση ενός κράτους που αποτελεί στρατηγικό εταίρο της ευρωπαϊκής ένωσης που διασφαλίζει την ενεργειακή ασφάλεια η τακτική αυτή απομακρύνει το αζερμπαϊτζάν από τον ευρωπαϊκό δρόμο. ποιο θα υποφεληθεί αν το αζερμπαϊτζάν κλείσει το δρόμο προς την πόρτα προ την ευρωπαϊκή ένωση προ τα πού θα στραπεί το αζερμπαϊτζάν ψηφίζω κατά του ψηφίσματο και υποστηρίζω την πρόταση να αναβληθεί η ψηφοφορία επί του συγκεκριμένου ψηφίσματο. Eh, και τώρα ο Επίτροπος Αβραμόπουλος για να κλείσει τη συζήτηση.

Το Αζερβαϊτζάν είναι τέρος στρατηγικής σημασίας για διάφορους ε, σημαντικούς στόχους, ε, ιδιαίτερα όσον αφορά την ασφάλεια ενέργειας και την περιφερειακή σταθερότητα. Η συνεργασία μας εντατικοποιήθηκε τα τελευταία χρόνια με βάση την ανατολική εταιρική σχέση και θα θέλαμε να δούμε αυτή τη σχέση να αναβημερεί και να αναπτύσσεται περαιτέρω επί τη βάση κοινών συμφερόντων και αξιών. Ωστόσο υπάρχουν σοβαρά θέματα στις σχέσεις μας που πρέπει να αντιμετωπιστούν ανοιχτά μεταξύ εταίρων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, παρακολουθεί στενά την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Αζερβαϊτζάν. Ε, συγκεκριμένα παρακολουθούμε τη δίκη του Ισλέιλα και του Καντήτιου Γιούνους καθώς και της ε, κυρίας Ισμαήλωβα όπως κάναμε νωρίτερα για τον κύριο Αζάροφ και τον ε, ε, ε, Αλίγεφ. Για να αναφέρω μόνο κάποιους από τους υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοσιογράφους στο Αζερβαϊτζάν. Αντιδράσαμε σε αυτές τις αρνητικές εξελίξεις με δηλώσεις μας, καθώς και σε άμεσες συζητήσεις σε υψηλότερο επίπεδο. Εξακολουθούμε να ζητούμε την απελευθέρωση με των ακτιβιστών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και ζητούμε δίκαιη δίκη. Θα θέλαμε το Αζερβαϊτζάν να ανταποκριθεί στι διεθνεί του δεσμεύσει ω μέλο του ΟΗΕ, του Συμβουλίου τη Ευρώπη και τη ΟΑΣΕ, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για την, ασφάλεια, την εξασφάλιση μάλλον τη ελευθερία, τη ελευθερία του ε, συνεταιρίζεσθε, την εφαρμογή του κράτου δικαίου μέσω ανεξαρτήτου δικαστικού σώματο ε, και με διαφάνεια. Δεν υποτιμούμε την ανεξαρτησία και την ε, ε, λειτουργία του ως σταθεροποιητή σε αυτή την ε, περιοχή. Θέλουμε να εξασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη σταθερότητα. Αυτό όμως θα γίνει μέσω της ελευθερίας των πολιτών να συμμετέχουν στην πολιτική συζήτηση. Γι' αυτό, δημοσιογράφους, γι αυτό οι δημοσιογράφοι θα πρέπει να μπορούν να ασκούν το λειτουργήμά τους ελεύθερα και να μένουμε περισσότερη δράση. Κατανοώ ότι οι αρχές ε, του Αζερβαϊτζάν ε, διερευνούν την πρόσφατη δολοφονία του δημοσιογράφου Μαλίγεφ. Εμεί προσπαθούμε ε, ε, να προωθήσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα και φαίνεται ότι έχει καλέ επαφέ με την κοινωνία των πολιτών στον Πακού. Η δική μα οικονομική βοήθεια είναι σημαντική σε αυτό το τομέα εφόσον στοχεύει στου πιο ευάλωτου τομεί και σημαίνει, κάνει διαφορά στι ε, ζωέ των ανθρώπων. Η αντιπροσωπεία μα επίση στηρίζει συγκεκριμένα ε, τους ε, υπερασπιστέ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα εξακολουθήσουμε να στηρίζουμε τις κοινέ μας αξίες και συμφέροντα στι διμερείς μα σχέσει καθώ και ε, στη, με βάση την Ανατολική Εταιρική Σχέση και ως μέλη και ιδίω του Συμβουλίου της Ευρώπης. Θέλουμε μια μακροπρόθεσμη επικοδομητική προσέγγιση που βασίζεται στη διάλογο τη δέσμευση και την εντατική χρήση των διπλωματικών οδών. Για να μπορέσουν οι σχέσεις μας να τοποθετηθούν επί νέων βάσεων, να αναπτυχθεί το δυναμικό, ε, θα ξεκινήσουμε διαρευνητικέ ε, συζητήσει με την Πακού την επόμενη εβδομάδα, ώστε να δημιουργηθούν νέε ευκαιρίε ε, για να συζητήσουμε το, με το Αζερβαϊτζάν και τα κοινά μα συμφέροντα και τι κοινέ μα δεσμεύσει. Έτσι να προσπαθήσουμε να μίξουμε το Αζερβαϊτζάν και να το, και, να το, να το παροτρύνουμε. Ωστόσο καταλαβαίνω ότι οι ορισμένοι βουλευτές δεν είναι ε, συμπαθούν την ιδέα της διαπραγμάτευσης με το Αζερβαϊτζάν από αυτές τις συνθήκες, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε κατά τη γνώμη μας αυτή την ευκαιρία για να επιδιώξουμε και στόχους ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αναπόσπαστο τμήμα των ευρύτερων μας σχέσεων. Το να χάσουμε αυτή την ευκαιρία δεν θα βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε τις ανησυχίες που όλοι έχουμε κοινέ εδώ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ Επίτροπε. Σας λέω ότι έχω λάβει 7 ε, προτάσεις ψηφίσματος μετά το πέρασε